yes, but I will give the word to him first, and then the rapporteur. Okay. okay. so, so, dear friends. Αγαπητοί φίλοι, ώρα είναι να ξεκινήσουμε. σχετικά με την ε, ομάδα εργασίας 3. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ε, πολίτες μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης. για τους ε, εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα, για την διακίνηση των ανθρώπων αλλά βέβαια με τον ίδιο τρόπο είναι πιο εύκολο για τους εγκληματίες να διακινούνται ελεύθερα διασυνοριακά και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών. Ε, Βεβαίω, ε, καταπολεμούμε αποτελεσματικά το διασυνοριακό έγκλημα και ελπίζουμε ότι θα διατηρήσουμε τις επιδόσεις αυτές γι' αυτό και πρέπει στην Ευρώπη να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην διευκρίνηση αυτών των εγκλημάτων. Και όπως είπαν και στην Ολομέλεια πολλοί, πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται μία ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης του εγκλήματος και της προστασίας των ε, ατόμων και των ιδιωτών. Πρέπει δηλαδή να ισοσκελίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ε, σχετικά με τις εγκληματίες και με τις διοκτικές αρχές και ε, να διευκρινίσουμε ακριβώς πώς θα γίνεται ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών, ποιες και πώς είναι οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται και πώς και τι πρέπει να διαφυλάξουμε για την ατομικότητα των πολιτών. Οι διοκτικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα αμοιβαία τις ε, τις του τους και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει αμοιβαία επιμόρφωση και ε, αυτά στα πλαίσια της ε, του προγράμματος Στοχόλμης. και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν και άλλες ιδέες που θα προκύψουν σήμερα. Επίσης ε, πόσο μπορεί να ενισχυθεί η δίωξη των υπόπτων για εγκληματικές πράξεις και υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία πρέπει να προασπίσουμε και ε, να διατυπώσουμε επίσης μακροπρόθεσμες προτάσεις στον τομέα αυτό. Όπως ε, γνωρίζετε υπάρχουν εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου άρα πρέπει να συσφίξουμε τη συνεργασία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα μας. Δεύτερον πρέπει να υπάρχει κοινή ε, δυνατότητα έρευνας και ανταλλαγή πληροφοριών και τρίτον πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την βαθμιαία προσέγγιση. Ε, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα εδώ και γι' αυτό θέλω καταρχήν να σας καλωσορίσω και να δώσω λόγο στην πρόεδρό μου κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντέβισον, συν πρόεδρε. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους εδώ για, αυτό, για αυτή την ομάδα εργασίας για την προστασία των πολιτών και την ευρωπαϊκή εσωτερική στρατηγική ασφαλείας δεν θα σχολιάσω το θέμα γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι δικές σας απόψεις και μία ανοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Σαν συντονιστής ή στην Επιτροπή Ελευθεριών ε, και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία και εγώ και η Επιτροπή μου ε, εις την συζήτηση των θεμάτων αυτών και στη συνεδρίαση που διοργανώθηκε σήμερα και ιδίως ε, σχετικά με τα θέματα αυτά. Είμαστε δηλαδή προσιλωμένοι στην εξέταση του θέματος αυτού και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των εθνικών εκπροσώπων διότι όντως όπως γνωρίζετε επειδή ε, εντός των επομένων ημερών θα ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν ε, διευρυμένο ρόλο σε αυτό το τομέα. Μήπως θα πρέπει να αναφερθώ λίγο στα θέματα ε, διαδικασιών. Θα δώσουμε τη δυνατότητα όσο δυνατόν σε περισσότερους να παρέμβουν. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το μπλε χαρτάκι που υπάρχει στο φάκελό σας για να μπορέσετε να εγγραφείτε ε, σαν στον κατάλογο των ομιλητών μας Ίσως ορισμένοι το αγνοούν αλλά όλοι πρέπει να ε, συμπληρώσετε αυτό το χαρτί και να μας το δώσετε για να μπορέσετε να εγγραφείτε στον κατάλογο των ομιλητών. Όταν θα ε, καλούμε έναν ομιλητή θα καλούμε και τον άμεσα ενδιαφερόμενο και τον επόμενο ομιλητή. Κατά τρόπον ώστε ο καθένας να ξέρει όταν επίκειται να λάβει τον λόγο. Προτού λοιπόν δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή στην, ε, στον κατάλογο επιτρέψτε μου καταρχήν να δώσω το λόγο στον εισηγητή της ομάδας εργασίας την κυρία ε, Κάρμεν Χερμόζαν Μπόνο που είναι πρόσωπος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ισπανίας και η οποία θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και θα ξεκινήσει έτσι την ανταλλαγή των απόψεων. Δίνω το λόγο λοιπόν στην ε, κυρία Χερμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Πολύ σύντομα, για να μην ε, χάσουμε χρόνο από τη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα πλαίσια αυτής της συνεδρίασης υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα είναι ζωτική σημασία. Αφενός έχουμε την ε, θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ε, συνέπεια αυτής της ε, θέσης σε ισχύ ο ρόλος που θα διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη συνέπεια και προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολούθησα την ε, συζήτηση στην Ολομέλεια. Παρουσιάστηκαν ε, διστάμενες απόψεις ε, για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά εδώ δεν θα ήθελα να ξεκινήσω κάποια συζήτηση και να προδικάσω οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσω όλα όσα έχουμε επιτύχει από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά, πλέον ε, εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις πολιτικές μετανάστευσης, να δούμε τι γίνεται με τις ε, μεταναστευτικές πολιτικές, όπως επίσης και με τις πολιτικές ασύλου έχουν ε, συσταθεί πολύ σημαντικοί ε, ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η Europol και ο Frontex και από εδώ και πέρα ε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα δώσει ουσιαστικά το ένασμα για τις νέες προκλήσεις οι οποίες θα τεθούν για το 2010 έως το 2014 στο χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Φυσικά η συνθήκη της Λισαβόνας και η θέση σε ισχύ της συνθήκης ε, θα ευνοήσει αυτές τις πολιτικές. Μία σύντομη σύνθεση. Οι βασικές προκλήσεις. Καταρχάς η ισορροπία, η πρόοδος και το να υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων με την ασφάλεια των ε, προσώπων πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα της ελευθερίας των ανθρώπων. Τα δικαιώματα του πολίτη θα είναι όλο και περισσότερο δεσμευτικά ε, στις ε, ευρωπαϊκές χώρες, όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ε, σημαντική προστασία ε, κατά των σημαντικών αδικημάτων όπως είναι η ξενοφοβία, ο ρατσισμός ε, και όλα όσα έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη και την συνεργασία σε μεταναστευτικές πολιτικές και πολιτικές ασύλου. Και τέλος να επισημάνω μία σειρά από προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να ζητήσουμε προληπτικά μέτρα και κάποιες διεκδικήσεις για νέα ή παλιά δικήματα τα οποία ε, σήμερα παρουσιάζονται με νέο πρόσωπο. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν μπορούμε να ρίξουμε τις άμυνές μας, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για τους πολίτες μας. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφέρω την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων, κυρίως ε, γυναικών και παιδιών, που ε, όχι μόνο είναι θύματα εμπορίου αλλά είναι και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι περισσότερες ε, γυναίκες ε, οι οποίες είναι οι τη σήμερα ημέρα είναι, έχουν προέλθει από εμπορία ανθρώπων. Υπάρχει επίσης το θέμα της παιδικής πορνογραφίας και της πειρατείας η οποία αφορά τα δικαιώματα των ε, δημιουργών καθώς επίσης και ε, τα παιδικά δικήματα που αφορούν τις οικογένειες, τα σχολεία και τις διάφορες οικογένειες. Τέλος, να σας πω ότι το πρόγραμμα που προτείνεται για τη Στοκχόλμη είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμενοποιηθούν ε, όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τις τροπολογίες που έγιναν. Και επειδή ακριβώς θα συμπέσει και με την Ισπανική Προεδρία, θα πρέπει ίσως να ετοιμάσουμε και ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο από όλη την έκταση του προγράμματος, το οποίο φυσικά θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διάφορα χρόνια, αυτό είναι λογικό, και ε, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, σταδιακά. Κάποια από τα στοιχεία που σας ανέφερα στην παρέμβασή μου θα πρέπει να περιλαμβάνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ερμοσίν Μπόνο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το ισπανικό σχέδιο δράσης, αυτό που θα υποβάλλετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ο κύριος Γκοντές είναι ο πρώτος μας ομιλητής. είναι βουλευτής από την Εθνοσυνέλευση της Σλοβενίας. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κύριος Γιόνκερ από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κύριος Γκόντες πάντως είναι ο πρώτος μας ομιλητής. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι το μήνυμα του προγράμματος της Στοκχόλμης είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι τα όρια μεταξύ της πραγματικής προστασίας ε, ε, των πολιτών της Ευρώπης ως ατόμων, των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό το όριο είναι πάρα πολύ λεπτό. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην το παρατραβήξουμε και να μεριμνήσουμε ώστε τα μέτρα που θα θεσπίσουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας να μην έχουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα η εξασφάλιση των Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να είναι ένα σημείο αφετηρίας για την εξασφάλιση και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει όμως να βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών της εξίσωσης. Για να έχουμε μια ασφαλή Ευρώπη θα πρέπει να ανακαλύψουμε τρόπους για να εγγυηθούμε αυτή την ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και την ιδιωτική σφαίρα, την ιδιωτική ζωή του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ως προς ότι η ασφάλεια είναι ένα συλλογικό αγαθό. Θα πρέπει να γίνει κάποια εναρμόνιση στα θέματα της ασφάλειας και να έχουμε και σχετική νομοθεσία. Η ευαισθητοποίηση του κοινού θα πρέπει να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Θα πρέπει να γίνει μια αφύπνιση και σε επίπεδο αρμόδιων αρχών, αλλά και σε επίπεδο απλού πολίτη. Θα πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει τις απειλές ε, που υφίσταται από τις διάφορες ε, μορφές του εγκλήματος, ε, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στη φάση της πρόληψης. Οπότε η επιτροπή μας, η προσοχή μας, συγγνώμη, καλό θα ήταν να εστιαστεί στα άτομα, στα ατομικά δικαιώματα, στις ατομικές ελευθερίες και προσοχή να μην να μην θυσιάσουμε στο βωμό της ασφάλειας τα ατομικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Γιόνκερ τώρα από την η κυρία Γιόνκερ μάλλον διορθώνει πρόεδρος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατόπιν θα λάβει το λόγο ο Ευρωβουλευτής Κάρλος Κοέλιο. Ευχαριστώ. Βεβαίως μιλώ από τη σκοπιά του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίωμα μας απασχολούν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέματα τα οποία συζητούνται επίσης στην Επιτροπή Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ε, ανέφερα διάφορα προγράμματα όπως συμφωνία για την ε, είσοδο, ε, προγράμματα επανεντάξεως κτλ. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι η Ευρώπη ποτέ δεν θα καταφέρει να επιστρέψει όλους τους παράνομους μετανάστες που έχουμε στην ε, Ευρώπη, κάπου 6,5 εκατομμύρια και ε, από την προοπτική του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ βασικό το πρόγραμμα της Στοχόλμης να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά με αυτούς τους παράτυπους μετανάστες και το πρόγραμμα της Στοχόλμης θα πρέπει να εξετάσει τι πρέπει να γίνει σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν μπορούν ή ε, δεν επιθυμούν να επιστρέψουν είναι ένα θέμα και νομικό και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο όμως ήθελα να... το οποίο είπα και στην Ολομέλεια, δηλαδή το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναφέρεται περισσότερο στη διαδικασία όσον αφορά τους μετανάστες και ε, όχι τις ε, διαδικασίες ε, οι οποίες άπτονται των, ε, των ροών μεταναστών. Οι άνθρωποι μας ενδιαφέρουν, όχι οι ροές τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Κάρλος Κοέλιο και μετά ο κύριος Άλμεν. Ο κύριος Κάρλος Κοέλιο μέρος της Επιτροπής Ελευθεριών. Έχω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό που συστήθηκε η ειδική ομάδα εργασίας για τα θέματα ασφάλειας. Κατά τη γνώμη μου, τα τρία σημεία, τρει συνιστώσει ε, του χώρου ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, η ελευθερία, και η δικαιοσύνη είναι αναπόσπαστα στοιχεία αυτού του τριγώνου. Δεν νοείται ο χώρο ε, ε, ελευθερία χωρί ασφάλεια γιατί η ελευθερία χωρίς ασφάλεια είναι αναρχία. Η ασφάλεια χωρίς ελευθερία είναι δικτατορία. Αλλά ούτε και η δικαιοσύνη νοείται χωρίς ασφάλεια και ελευθερία. Η ασφάλεια λοιπόν αποτελεί ένα στοιχείο, έναν απόσπαστο στοιχείο της ε, ελευθερίας και μία εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση της δικαιοσύνης. Μερικές φορές αντιμετωπίζεται η ασφάλεια συγγνώμη, ως εχθρός της ελευθερίας. Νομίζω ότι είναι σαθρό αυτό το επιχείρημα, πολύ περίπλοκη προσπάθεια να χειραγωγηθεί. Όπως είπα και στην Ολομέλεια, πέραν των αρχών και των αξιών, δεν θα πρέπει να μελούμε και την αρχή της αποτελεσματικότητας. Και εκεί είναι που χωλαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Στο χώρο Σέγγεν, το πιο σημαντικό σημείο είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εγγύηση ότι ένα πολίτη ε, τρίτη χώρα εισέρχεται στην Πορτογαλία, ο Πορτογάλος ακριτοφύλακας θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες πληροφορίες από όλες τις υπόλοιπες χώρες μέλη, αν θα πρέπει να επιτρέψει την είσοδο σε αυτόν τον πολίτη τη χώρας ή θα πρέπει να τον παρακολουθήσει. Αυτό το νόημα έχει ο χώρο Σέγγεν και η πρώτη γενιά του συστήματος Σέγγεν. Η δεύτερη γενιά του συστήματος πληροφόρου Σέγγεν ε, προσθέτει μια αξία γιατί χάρη στα βιομετρικά στοιχεία απαλλάσσεται από τον κίνδυνο να λάβει υπόψη κάποια πλαστά έγγραφα. Επίσης ε, κάνει τη διάκριση μεταξύ μιας κλοπής που έγινε απλώς για να κλαπεί ένα αυτοκίνητο ή μιας κλοπής που είναι τμήμα ενός κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης θα πρέπει, το σύστημα θα πρέπει να έχει τεθεί σε το 2007, αλλά έχουμε φτάσει το 2009 και κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το 2012 δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ. Γι' αυτό και είπα στην εναρτήρια μας συνεδρίαση, πριν προσθέσουμε νέους στόχους και νέες προκλήσεις, καλό θα ήταν να, ε, να περάσουμε ένα τεστ αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας. Εκεί να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Γιατί εκεί έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, ώστε να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα πρώτα, πρώτα πριν περάσουμε στα επόμενα μέτρα. Ευχαριστώ, Κάρλος. Το λόγο έχει ο κύριος Άλμπερτ, που είναι μέλος της Γερουσίας της Ρουμανίας και μετά θα ακούσουμε ένα εκπρόσωπο της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλησπέρα κύριε και κύριοι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δώσαμε τη δέωσα προσοχή στην Ολομέλεια για τα όσα θα πρέπει να προσέξουμε, τις προκλήσεις που μας περιμένουν για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως είπαν πολλοί από τους προλαλήσαντες και εδώ αλλά και στην Ολομέλεια, η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την ευημερία και την ελευθερία. Η πραγματικότητα σήμερα Μα βρίσκει αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλες ε, προκλήσεις. Η οικονομική κρίση, οι κλιματικές αλλαγές, ε, ε, θέματα μετανάστευση και όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προασπίσουν τα κοινά του συμφέροντα. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έχει προχωρήσει και είναι πλέον κάτι το οποίο είναι τμήμα των κοινωνιών μας. Το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθεί να απειλεί τις κοινότητές μας ε, με το εμπόριο ναρκωτικών ε, και για να μπορέσουμε να... και άλλα εγκλήματα και για να μπορέσουμε να ε, να καταπολεμήσουμε τα θέματα αυτά θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εξαρθρώσουμε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αστυνομική και δικαστική συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βρίσκουν καταφύγιο οι εγκληματίες ε, σε ευρωπαϊκά εδάφη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία ε, μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο πληροφοριών και να πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα και σε έγγραφα για τις διάφορες ε, υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών. Και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωμανία έχει μια συγκεκριμένη πρόκληση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Για να μπορέσει να συνεργαστεί λοιπόν σε θέματα ασφάλειας θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους γείτονε μας. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία και να μπορέσουμε να έχουμε και μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέσα, ε, συμφωνίες ε, συνεργασίας και εταιρική σχέσης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πάγιες πολιτικές ε, και σε επίπεδο πολιτικό με τους εταίρους μας από την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άλμπερτ. Να θυμίσω ο μόλις έφτασε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριος Σταύρος Λαμπρινίδης εδώ και σας ευχαριστώ επίσης να σέβεστε τα, την προθεσμία τριών λεπτών. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά η κυρία Απτουλά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε ε, Πρόεδρε, το 1992 καταρτήσαμε την ενιαία αγορά, αλλά ξεχάσαμε τους ε, εγκληματίες οι οποίοι αλωνίζουν την Ευρώπη και πρέπει τώρα να μπορέσουμε να βρούμε ένα σύστημα για να τους ε, ε, διώξουμε και να τους συλλάβουμε και γι' αυτό θα πρέπει να συντονιστεί η εργασία των αστυνομιών της Ευρώπης. Στην έκθεση είδαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για να ανταλλάξουν πληροφορίες ε, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών αρχών και της Europol, ιδίω όσον αφορά τις πληροφορίες ασφαλείας και τις εμπιστευτικές και στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι περισσότεροι νόμοι δεν ξέρουν ξένες γλώσσες και όταν εξετάζουν έναν ύποπτο από την κεντρική Ευρώπη του μιλούν αγγλικά και ελπίζουν ότι θα απαντήσει. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις να είναι στο ίδιο επίπεδο για να μπορέσει και η Ευρωπόλ να λειτουργήσει σωστά. Ε, επίσης ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της χρειάζεται βελτίωση και η Europol και η Eurojust ε, που είναι τόσο βασικό να συνεργαστούν παρόλο που βρίσκονται στη Χάγη δεν ε, ε, βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και όταν τους επισκεφθήκαμε είδαμε ότι αν ήταν σε ένα κτίριο θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική αστυνόμευση και ε, να μπορέσουν να συλλάβουν τους ε, εγκληματίες για να τους αναλάβει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκτιμά τις ε, έρευνες τις οποίες κάνετε, τις επισκέψεις, τις ανταλλαγές με ευρωβουλευτές. Είναι μία άσκηση που εκτιμούμε πάρα πολύ. Τώρα η κυρία Ζήση Ραδούλα από το Ελληνικό Ελληνικό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια ο κύριος Λίνμπλατ Γκόραν. Ε, είναι σαφές ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι η πρόκληση και η πρόσκληση, η ισορροπία και η συμβατότητα όπως ακούστηκε εδώ μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, της Νέας Χάρτας, αλλά βεβαίως και της ασφάλειας που είναι κοινωνικό αγαθό. Μέσα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες της ένωσης προϋποθέτει την αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικής δραστηριότητας και κυρίως αυτών που στρέφονται κατά των σημαντικότερων αγαθών των πολιτών όπως είναι η ζωή η σωματική ακεραιότητα η περιουσία. πρέπει λοιπόν παράλληλα με όλο αυτό που συζητάμε να υπάρξει και ένας ισχυρός μηχανισμός πολιτικής προστασίας τι επιβάλλεται τώρα κατά την άποψή μας μια συστηματική και συντονισμένη αντιμετώπιση όλων αυτών και θα σταθώ στα σημεία τα εξή πρόβλεψη πρόληψη διάγνωση κάθε νέας απειλής και αποτροπή κυρίως στις περιοχές που υπάρχουν διασυνοριακά και υπερεθνικά ζητήματα ε, είναι απαραίτητη αυτή η πρόληψη και βεβαίως τα μέτρα ε, κατά όλων αυτών των φαινομένων πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενίσχυση και θωράκιση των δεσμεύσεων των πολιτικών αθενών αλλά ενίσχυση και αξιοποίηση των θεσμικών οργάνων της ευρωπαϊκής ένωσης συνεργασία τους με διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως χρειάζεται η βελτίωση του επίπεδου της συνεργασίας των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ε, των κρατών μελών πάντα με την αποφασιστική συμβολή της europol και της eurojust. πιστεύουμε ότι η καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας θα φέρει πάλι καλύτερα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδιορίσει τις βασικές ζώνες προτεραιότητας που κατά τεκμήριο αποτελούν τις ε, γενουσεριές αιτίες απειλής πρέπει λοιπόν να αναπτύξει επαφές με τις χώρες της εν λόγω περιοχές με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχους αλλά και χρησιμοποιώντας τα θεσμικά εργαλεία και τα κατάλληλα μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής. πιστεύουμε ότι η ειρήνη η συνεργασία και η πρόοδος σε αυτό το τομέα θα δώσει πραγματικά μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική τα καλύτερα αποτελέσματα. σε σχέση τώρα με την τρομοκρατία και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ διευκολύνουν τι δραστηριότητε αυτέ. Χρειάζεται εδώ, όπω πολύ σωστά υπόθηκε, μια ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, αλλά και ενίσχυση των πολιτικών για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Χρειάζεται να προβλεφθούν ε, και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Στοκχόλμη η πρόβλεψη για τη χρήση νέων τεχνολογιών, να αξιοποιηθεί δηλαδή όλη η εμπειρία που έχουμε, υπό την προπόθεση πάντα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφύλαξης του απορρίτου των δεδομένων. Η αποκέντρωση των δομών της Frontex και η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της θα φέρουν και, αυτά πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Υποστηρίζουμε εμείς παράλληλα και τη διεύρυνση ε, αρμοδιοτήτων αλλά και συγκρότησης ενός περιφερειακού βραχίωνα της Frontex στη Μεσόγειο θάλασσα και στην ευρωμεσογειακή ε, τελικά ε, λεκάνη και συνεργασία. Τέλος, αναφερόμενοι στη διευκόλυνση πρόσβασης στη δικαιοσύνη από τους Ευρωπαίους πολίτες, θεωρούμε απαραίτητη την υιοθέτηση δικονομικών δικαιωμάτων, διότι έτσι θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πιστεύουμε ότι η προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί παροχή εγγυήσεων πρόσβασης σε υπηρεσίες διερμηνίας και μετάφρασης στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας, καθώς επίσης και η παροχή πληροφοριών και η δικαστική συνδρομή. Θα δώσουμε με τη θωράκιση αυτή, με τα μέτρα τις δράσεις, τη συνεργασία και τον πυλώνα της αλληλεγγύης που πρέπει να ενισχυθεί, στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης το ξεκάθαρο μήνυμα του προγράμματος της Οκχόλμης, το ξεκάθαρο μήνυμα του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη θεμελιώδη ελευθερία, στην αρχή του κράτους δικαίου, σε αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ και όλοι με την πιο καλή μας πρόθεση θέλουμε να ενισχύσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Πάντως υπερβήκατε λίγο το χρονικό σας όριο, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε που δεν τόλμησα να σας διακόψω. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λίμπλαντ Κόραν και θέλω παρακαλώ τους λοιπούς ομιλητές να μην ξεπεράσουν το τρίλεπτο και μετά η κυρία Μούλτι Ρωσάνα. Ο κύριος Λίμπλαντ Γκόραν προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άλλωστε είμαι και πρόεδρος ε, της, Επιτροπής Πολιτικών ε, ε, θεμάτων και αναπληρωματικό μέλος ε, στην Επιτροπή Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε κάποιες τροπολογίες ε, που θα καταθέσουμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και ευελπιστούμε ότι θα τις μελετήσουν οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευελπιστούμε ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν και τη σχετική συζήτηση θα τις εγκρίνουν. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ας μην ξεχνούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, ασχολούμαι ιδιαίτερα με θέματα δημοκρατίας, ε, κράτους δικαίου και ελευθερίας και είμαι υπέρ της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα βέβαια της μετανάστευσης. Να μην ασχοληθούμε δηλαδή μόνο με τους ε, νόμιμους μετανάστες, αλλά και με τους λαθρομετανάστευση. Δεν θα πρέπει να μιλούμε για παράνομη μετανάστευση, γιατί όταν λέμε το παράνομος δίνουμε λάθος μήνυμα στο σύστημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν τίποτα παράνομο. Ε, προσπάθησαν να γλιτώσουν από μια οικονομική δυσπραγία, από ένα πόλεμο ή από μια δικτατορία, από την κατάσταση στη χώρα τους και δεν πηγαίνουν ε, προς ένα μέρος, αλλά φεύγουν ε, από κάποιο μέρο ζητώντα προστασία. Δεν έκαναν τίποτα παράνομο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να του προστατεύσουμε. Επίση, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ε, και οδοντιατρική περίθαλψη. Ε, γιατί όταν ε, δεν συνεδριάζω στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, ασκώ. Έχω ιατρείο, οδοντιατρείο και βλέπω τέτοιου ανθρώπου. Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι φυλακισμένοι. Και μάλιστα επειδή για 20 χρόνια υπηρετούσα σε φυλακή και φρόντιζα τα δόντια φυλακισμένων, βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Παρόλο που δεν έχουν κάνει τίποτα παράνομο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσουν τη φωνή του και να προστατεύσουν αυτού που περισσότερο το έχουν ανάγκη. Η κυρία Μόλντι Ρωσάνα από την Ιταλική Γερουσία και μετά ο Ζανζάκ Καμπενιστή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή αυτής της ομάδας εργασίας ε, που αφορά στην προστασία των πολιτών στην, ε, στον οργανισμό της Frontex. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια αποτελεσματική απάντηση με συνολική προσέγγιση στα θέματα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες να ε, χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές και να διασφαλίσουν την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων ε, και την ε, καταπολέμηση της ε, κακομεταχείρισης των ανθρώπων και την ανάγκη διαχείρισης πολύ ισχυρών μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να υπάρχει λειτουργική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω του οργανισμού της Frontex θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, περισσότερες δομές, σε τελευταία ανάλυση και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την διεξαγωγή των ε, δραστηριοτήτων της θα πρέπει να υπάρχουν ε, δευτερεύουσες έδρες ή κάποια ειδικά γραφεία της Frontex ε, σε περιοχές οι οποίες ε, χρειάζονται ιδιαίτερες επιχειρησιακές ικανότητες σε θέματα διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως στη λεκάνη της Μεσογείου. Επίσης θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετανάστευσης ο οποίος θα προκύψει από τις κοινέ προσπάθειες όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν, να τις αρμοδιότητες στο το κόστος, τις πολιτικές επιπτώσεις και τα συνέπειες της μετανάστευσης, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν κυρίως τις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία οπισθοχώρηση στα θέματα αυτά σε σχέση με τα όσα έχουν καθοριστεί σε όλες τις συνεδριάσεις που έχουν γίνει από τον Οκτώβριο του 2008 και τούδε και τέλος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης και 30ης Οκτωβρίου είναι ζωτική σημασία για την ε, ε, προάσπιση των συνόρων στα νότια της Ευρώπης να υπάρχει συντονισμός με τις χώρες της Μεσογείου. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ε, για τη Λιβύη επί παραδείγματι ότι η κυρία Φεραίρο Βάλνερ είχε αναλάβει συγκεκριμένε δεσμεύσει με τη Λιβύη για τη χρηματοδότηση ενό δορυφορικού συστήματο ε, παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών που προέρχονται από τα νότια Σύρια, ε, σύνορα τη Λιβύη, το οποίο δεν είχε καμία συνέχεια. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω αφορά την ανάπτυξη πολιτικών ε, για την ε, αντιμετώπιση των εγκληματικών δράσεων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση πλαίσιο και να, ρυθμούν, ε, να ληφθούν μέτρα τα οποία θα έχουν και ποινικέ συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα πηγαίνει στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη. Α, συγγνώμη, πριν από τον κύριο Λαμπρινίδη, ο λόγο στον κύριο Μπενίστη, τον οποίο είχα ήδη αναγγείλει και μετά θα λάβει το λόγο ο κύριο Λαμπρινίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να παρέμβω και να πω ότι όλοι πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουν για μια ανταλλαγή ε, πληροφοριών διασυνοριακά και τα κράτη-μέλη να ε, επιτρέψουν αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένες εθνικές βάσεις δεδομένων. Είτε πρόκειται για ε, τους φακέλους του ADN διότι η συμφωνία PROM υπερβαίνει επαναλαμβάνει την συμφωνία πλαίσιο του 2008 και εκεί επιτρέπεται η μεταβίβαση πληροφοριών που υπάρχουν στις ε, αστυνομικές και δικαστικές ε, εθνικές ε, καταστάσεις χωρίς όμως να είναι αυτοματιοποιημένη, δηλαδή άμεση. Στα πλαίσια της συμφωνίας ΠΡΟΜ οι πληροφορίες μεταβιβάζονται μέχρι, μέσω του συστήματος ΤΕΣΤΑ 2 παραμένει ανώνυμη το σύστημα και μόνο σε περίπτωση ε, ταυτίσεως μπορούν να ε, δοθούν τα προσωπικά στοιχεία για το ADN ή για ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Διαφορετικά οι Γάλλοι θα έχουν δυνατότητα να έχουν μόνο το αντίγραφο της βάσης δεδομένων αυτής επί τη ευκαιρία της συμφωνίας των Υπουργών Δικαιοσύνης στη Δρέσδη το 2005 όπου παρουσιάστηκαν η συνεργασία των γερμανικών και αυστριακών αρχών στο πλαίσιο αυτό και βρεθήκαν πάνω από 500 50 σε χίλιες εκ των οποίων 30 για εγκλήματα και ένας αριθμός επίσης για σεξουαλικά εγκλήματα. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές της ΕΟΚ να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους βάση, στις δικές τους βάσεις δεδομένων και να υπάρχει μία διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κατασταλτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι μόνο έτσι θα μπορέσει κανείς και να προστατεύσει τα δεδομένα και να υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λαμπρινίδης. Ευρωβουλευτές ε, το ε, μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας και μετά ο κύριος Πάουελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα χαρά σας βλέπω εδώ, διότι όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα είναι θέματα συναποφάσεως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υπόκεινται με τη συνθήκη της Λισαβόνας και σε εθνικό έλεγχο. Ε, με την κυρία ζήσει Ζήση Αβδούλα είχα την δυνατότητα να συζητήσω το θέμα αυτό διότι είναι και η υπεύθυνη για την αρμόδια επιτροπή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τρόπο ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα εφόσον θεωρείτε ότι τα κοινοβούλια στις χώρες σας χρειάζονται αυτές ε, τις δυνατότητες να συζητήσετε ε, μεταξύ των εθνικών βουλευτών σας και των ευρωβουλευτών σας διότι ε, διαφορετικά το σύστημα θα είναι άχρηστο. Εμείς θέλουμε από κοινού να μπορούμε να εξασκούμε τις ε, δημοκρατικές μας δυνατότητες προβλέπουμε ότι το ε, διαδίκτυο θα είναι το επόμενο πεδίο μάχης μεταξύ ασφαλείας ε, και ανταλλαγής πληροφοριών διότι ε, ναι μεν οι διοκτικές αρχές θέλουν να έχουν ε, την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στα στοιχεία που χρειάζονται και πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα μπορέσει το διαδίκτυο και να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμα του εκφράζεστε, το δικαίωμα του έρχεστε και από την άλλη πλευρά να μπορεί να ελέγχεται για την σύλληψη των μελλοντικών εγκληματιών. Αυτό το Κοινοβούλιο και αυτό το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή Προ δύο εβδομάδων συνεφώνησαν το τηλεπικοινωνιακό πακέτο, ιδίως για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οπότε συζητήθηκε να περιοριστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και εμείς αποφασίσαμε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα όπως και τα άλλα. Άρα οι υπερβονικές ποινές ε, για αυτούς τους λόγους δεν πρέπει να προωθηθούν ασκηθούν εκτός ε, αν υπάρχει εκ προημίου έλεγχος από δικαστήριο και εξουσιοδότηση από το δικαστήριο. Αυτά ήθελα να σας πω και θα ήθελα να το τονίσω. Και ο άλλος λόγος αγαπητοί φίλοι, εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση κύριε Πρόεδρε, σκεφτείτε το εξής. Σε κανένα κράτος η αστυνομία δεν μπορεί να ανοίξει ένα γράμμα το οποίο στέλνουμε στο ταχυδρομείο για να το διαβάσει και να πει αν αυτό που γράφω εγώ στον Κάρλος Κοέλιο ας πούμε μπορεί να περιέχει γλώσσα από τα οποία απορρέει ότι μπορεί να είμαι τρομοκράτης. Ε, είναι πολύ πιο πιο εύκολο όμως να ελέγξει κανείς ε, τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Εάν δεν ε, ε, επιτρέπουμε λοιπόν στην αστυνομία ή σε μια ιδιωτική εταιρεία να ανοίξει τα γράμματα στο ταχυδρομείο, γιατί θα έπρεπε η αστυνομία ή οι ιδιωτικές εταιρείες να ελέγχουν τα προσωπικά μας μηνύματα στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά μηνύματα ε, πολλοί από εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τομείς όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την νομοθεσία. Το πρώτο θέμα είναι ε, για την μετανάστευση που είναι ένα εθνικό θέμα αλλά όταν αποτυγχάνει η ενσωμάτωση τότε πρέπει να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή και το πιο βασικό είναι είναι όλη, όλα τα θέματα της ε, συνθήκης της Λισαβόνας όπου στη Γαλλία και στην Ολλανδία ε, δεν ε, εστιάστηκε η προσοχή στα δικαιώματα των Γάλλων ή των Ολλανδών αλλά το εάν η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αν θα μπορούσαν έτσι να μεταναστεύουν ανεξέλεγκτα μουσουλμάνοι. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και όμως έγινε. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης είναι κάτι που πρέπει να γίνει βάσει μια στρατηγική σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Δεν πρέπει να λέμε ότι έχουμε βέλτιστες πρακτικές αν δεν μπορούμε να τις ανταλλάξουμε. Δεύτερον, υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές, διότι ορισμένες χώρες για γεωγραφικούς λόγους έχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ε, μεταναστών ε, είτε επισήμων είτε ανεπισήμων όπως η Μάλτα, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, ακόμη και η Ισπανία. Υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες ροές αλλά όπου η υπόλοιπη Ευρώπη τις αντιμετωπίζει λέγοντας ότι αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ολονών μας, όχι μόνο για να ελέγχουμε τα σύνορά μας για θέματα συνόμευσης, αλλά και για λόγους ανθρωπιστικούς και ανθρώπινους. Να μπορούν τα άτομα αυτά είτε να εισέλθουν ε, στην κοινωνία μας, είτε να επιστρέψουν στην ε, πατρίδα τους εάν μπορούν. Μετά, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν έχω δει το ψήφισμα και τις τροπολογίες τις οποίες προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα ήθελα να τις δω, αλλά προτού προτείνεται νέα μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Για προσπαθήστε να δείτε αν τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν ε, εφαρμόζονται και ε, γίνονται σεβαστά διότι δεν αρκεί να έχουμε νέα μέτρα για να πιάσουμε τον κακό αλλά για να εξετάσουμε πώς θα έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά διότι τώρα έχουμε τόσες συνθήκες, ε, Schengen 2, ΠΡΟΜ, Eurodac, SWIFT, οι διαπραγματεύσεις SWIFT ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα τραπεζικά στοιχεία. Είναι θέματα τα οποία ακόμη δεν εφαρμόζονται ενιαία και προτού αξιολογήσουν πώς αλληλεπηρεάζονται ήδη μιλάμε για νέα μέτρα. Αγαπητοί φίλοι, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου για να μπορέσουμε να έχουμε μία σοφή πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους τρομοκράτες να διακινούνται ανεξέλεγκτα αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και ποια μέτρα είναι αποτελεσματικά διότι διαφορετικά φοβόμενοι ε, νέα εγκλήματα θα έχουμε νέα μέτρα που θα περιορίσουν τα δικαιώματα αντί να πιάνουν τους εγκληματίες. Ε, ευχαριστώ που μου δώσατε τον χρόνο να μπορέσω να εκφραστώ. Βλέπω όμως ότι κύριε Λαμπρινίδη υποφεληθήκατε από το λάθος μας και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιάν Μπάουερ από την Τσεχία και μετά ο Τόλι Ταπάνη από τη Φιλανδία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που μας δίνετε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Έχω μερικές παρατηρήσεις. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλη τη συζήτηση και στην Ολομέλεια και εδώ και νομίζω ότι η, η λέξη που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι κράτος δικαίου και δικαίωμα. Δικαιώματα παιδιών, δικαιώματα ε, προσφύγων. Δεν ακούμε όμως ε, αρκετά συχνά τον όρο υποχρέωση και ευθύνη. Όλα για δικαιώματα μιλούμε, αλλά για ευθύνε και υποχρεώσει ε, λέμε ελάχιστα. Ενώ μία κοινωνία μπορεί να είναι επιτυχής όταν σέβεται τα δικαιώματα, αλλά όταν τηρεί και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Έχω και ένα σχόλιο ε, που είναι προσωπικό μου βίωμα, γιατί το μισό της ζωής μου το πέρασε υπό ένα πολιτερχικό καθεστώς και όσο βρισκόμουν στο ζυγό αυτού του καθεστώτος σκεφτόμουν τι είδου κριτήρια γίνονται δεκτά για τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες σε δημοκρατικές χώρες. Ακόμη για πρόσφυγες ε, και μετανάστες ακόμη και από χώρες της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα είμαι πια Μέλο αυτή τη νέα διευρυμένη Ευρώπη και μπορώ να συμβάλλω και εγώ για τη διαμόρφωση αυτών των κριτηρίων αποδοχή των μεταναστών γιατί όλοι συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κοινά μέτρα σεβόμενοι τις κοινέ μας αξίες. Δεν θα ήθελα να κλειστούμε, να ορθώσουμε τείχους και να είμαστε αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε και πολλές συζητήσεις για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πολλοί πολιτικοί έχουν τόσο υπέρμετρες φιλοδοξίες που θα χρειάζονταν δύο κοινοτικού προϋπολογισμούς για να τις υλοποιήσουν. Κάτι που εκνευρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες. Η υπερβολική φιλοδοξία τους εκνευρίζει όσο και η απόλυτη έλλειψη φιλοδοξίας. Θα πρέπει να βρούμε το μέτρο μεταξύ των δύο. Και κάτι άλλο για το οργανωμένο έγκλημα. Πολύ συχνά οι εγκληματίες ε, προπορεύονται είναι ένα βήμα πριν από εμά και είναι σωστό να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και διασύνδεση. Α μην ξεχνούμε ότι αν ενισχύσουμε αυτή τη διασύνδεση, πολύ πιθανόν, αν δεν ε, τονίσουμε την προστασία των δεδομένων, να εκμεταλλευτούν αυτή τη διασύνδεση και την ανταλλαγή πληροφοριών πρώτα απ' όλα οι εγκληματίε. Ο κύριος από τη Φιλανδία έχει το λόγο και μετά εκπρόσωπος του Βελγίου. Σας ευχαριστώ έλαβα το λόγο και στην Ολομέλεια και εκεί τόνιζα, τόνισα την ανάγκη μιας εναρμονισμένης πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όμως τι σημαίνει μια τέτοια κοινή πολιτική ασύλου. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει φυσικά σωστή διαχείριση και έλεγχο των συνόρων και αυτό θα μας το εξασφαλίσει ο οργανισμός Frontex. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη Frontex για να αναλάβει αυτόν τον ε, ενισχυμένο ρόλο. Βέβαια δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από τη Frontex. Έχουμε και πρόβλημα με τούντες ασύλο που έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τα κυκλώματα οργανωμένου έγκληματος. Πολλές φορές ε, εγκληματίες διακινούν λαθρομετανάστες και μάλιστα ζητούν αστρονομικά ποσά για να φέρουν αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το κάνουν παράνομα μέσα στη νύχτα με δεινές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια εναρμονισμένη πολιτική ασύλου που θα σέβεται φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλουμε ε, αυτοί οι λαθρομετανάστες να εισέρχονται στην Ευρώπη και να μετατρέπονται σε παράνομο εργατικό δυναμικό από με, λαθρομετανάστες να γίνονται μετά λαθροεργάτες. Θέλουμε παρόμοιες διαδικασίες ε, επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου. Μια εναρμονισμένη πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα την αστυνομία, πιστεύω ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι καλός προς την ουσία του και τις βασικές του γραμμές. Χρειαζόμαστε τη σωστή στρατηγική για να επεξεργαστούμε αιτήσει ασύλου και φυσικά χρειαζόμαστε και σωστή στρατηγική απασχόληση αλλά και τη χρήση των νέων τεχνολογιών που θα εξυπηρετούν και την ασφάλεια των πολιτών μας. Γι' αυτό φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων της Ευρώπης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική συνεργασία και η Φιλανδία είχε αρκετές προτάσεις γι' αυτό και μάλιστα υπάρχει και ένα πειραματικό ε, πρόγραμμα συνεργασίας ε, που προτάθηκε από τη Σουηδική Προεδρία για την τελωνιακή συνεργασία και την αστυνομική συνεργασία. Θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση της απειλής που σημαίνει για μας το οργανωμένο έγκλημα. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους αστυνομικούς ε, να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. Επίσης χρειαζόμαστε και περιφερειακή συνεργασία με τους γειτονές μας, για παράδειγμα τη Ρωσία. Το λόγο έχει η κυρία Ζακλίν Ένα από το Βέλιο και μετά ο κύριος Κρίστοφ Χάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνική. Θα ασχοληθώ με τρία σημεία. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την αστυνομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνεται πολλής λόγος για την αστυνομική συνεργασία με τις ε, γειτονικέ χώρες του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά πρώτα θα πρέπει να ενισχύσουμε την αστυνομική συνεργασία εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Εγώ κατάγομαι από την περιοχή του ΕΝΟ, που είναι όμορη της Γαλλίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα των ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε καν τα μέσα να αντιμετωπίσουμε ε, διασυνοριακό έγκλημα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Βρισκόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό χώρο και άρα είμαστε αρκετά απαλλαγμένοι από τους πολέμους και την απειλή στην ανθρώπινη ζωή, αλλά έχουμε πολλούς πρόσφυγες από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, έχουμε μια τοπική πρωτοβουλία υποδοχής από ε, υπηκόους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που επικαλούνται πολιτικούς λόγους ε, και ζητούν πολιτικό άσυλο, κάτι που είναι αδιανόητο για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για το Φιλελεύθερο Κόμμα του Βελγίου έχει σημασία η οικονομική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών, ειδικά για, τη, για τα επαγγέλματα που υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για να καλυφθούν αυτές οι κενές θέσεις ε, εργασίας ή τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σπάνι να καλυφθούν εσωτερικά από Ευρωπαίους πολίτες και να μην έρχονται υπήκοοι τρίτων χωρών να παίρνουν τις θέσεις ε, Ευρωπαίων πολιτών. Και η Γαλλία πρότεινε παρόμοιε πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθεί μια οικονομική μετανάστευση έσω κοινοτική ώστε να καλυφθούν ε, θέσεις σε επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σπάνι. Ευχαριστώ ο κύριος Κριστον Χάγκεν από το Αυστριακό Κοινοβούλιο τώρα και μετά ο κύριος Σούφς από το Βέλγιο που είναι και ο τελευταίος ομιλητής που έχω στον κατάλογό μου εκτός και αν κάποιος άλλος θέλει να εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλωτών Αλλιώς θα κλείσει ο κατάλογος. Παρακαλώ λοιπόν αν θέλετε να μιλήσετε να το πείτε τώρα. Ο λόγος πηγαίνει στον κύριο Χάγκεν. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αστυνομική συνεργασία και ο συντονισμός στην Ευρώπη μου φαίνεται ένα πολύ βασικό στοιχείο, ιδίως διασυνοριακά η Αυστρία εδώ ακολουθεί μία άλλη κατεύθυνση διότι έχουμε ήδη εφαρμόσει την ε, διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με τα γειτονικά μας κράτη. Από το 2008 έχουμε ε, έρθει σε επαφή με τους ε, υπαλλήλους οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα νομικά και άλλα και έτσι την Πέμπτη στο Εθνικό μας θα αποφασίσουμε ότι οι ξένοι αστυνομικοί θα έχουν ενισχυμένα δικαιώματα να παρέμβουν στην Αυστρία ε, και αυτό είναι ένα πρώτο βασικό βήμα και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει και τα άλλα εθνικά κράτη να μπορέσουν να δώσουν δυνατότητες σε όλες τις εθνικές αστυνομικές μονάδες στην Ευρώπη για να μπορέσουν να συνεργάζονται και να έχουν ε, ε, συνεργασία και με τις ξένες δυνάμεις. Το σύστημα ε, πληροφοριών Schengen SIS 2 δεν ισχύει ακόμη δεν λειτουργεί ακόμη και πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια επιτάχυση ε, των προσπαθειών διότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Θα είμαι σύντομος διότι έχουμε λίγο χρόνο. Το άσυλο όμως είναι για μένα επίσης πολύ σημαντικό γιατί ελέγχθη ότι κράτη όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και άλλα είναι πολύ επιβεβαρημένα αλλά η Αυστρία που είναι στη μέση Ευρώπης, στο κέντρο της Ευρώπης Έχω, έχει ήδη 18.000 αιτήσει ε, ασύλου και νομίζω το πρόβλημα είναι διευρωπαϊκό και θα έπρεπε όλα τα κράτη να βοηθηθούν. Το δικαίωμα ασύλου είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να περιληφθεί στις, στα θέματα που επεξεργάζεται η Ευρώπη γενικότερα και ε, όσον αφορά τις χώρες ε, όπου υπάρχουν εξωτερικά σύνορα της ε, Ένωσης θα πρέπει να έχουν ενισχυμένη παρουσία της Frontex και για τις νέες χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν πολύ καλά συστήματα να τύχουν ως Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποβλέποντας σε μία βελτίωση, δηλαδή ε, να διατεθούν στα κράτη αυτά και χρηματικοί και γενικότεροι πόροι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν καλύτερα σε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο τελευταίος ομιλητής είναι ο Μπέρτ Σούφς από το Βελγικό Κοινοβούλιο και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα της μετανάστευσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι συχνά η εισαγωγή της μετανάστευσης σημαίνει εισαγωγή ένδυας αλλά και εργατικό δυναμικό ε, το οποίο χάνεται από τις χώρες ε, προέλευσης. Αυτά τα άτομα πρέπει να τα υιοθετούμε, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει πρωτίστως να σκεφτεί πώς μπορεί να τους επαναπατρίσει ε, στις χώρες τους με αποτελεσματικό τρόπο και προφανώς δίνοντας και αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες προέλευσης, κυρίως στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν σειράξεις. Σαφώς υπάρχουν ε, άνθρωποι καλή την προθέση, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, λιγότερο καλές προθέσεις. Επί παραδείγματι, εξακολουθεί να υπάρχει ε, εμπόριο υλικού το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βόμβας ή να καταλήξει στα χέρια τρομοκρατών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία ε, σταθερή δομή δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχουν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα αλλά δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ισχύει και για τις ε, χώρες μας, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια ανθρώπινη Ευρώπη η οποία θα σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν και ε, ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι ο ρόλος της ε, Europol και της Eurojust, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία, διότι στο τέλος θα πρέπει να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κυριαρχία των κρατών μελών και εξετάζοντας τους ενδεχόμενους κινδύνους ε, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να έχουμε ένα κέντρο ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα του ελέγχου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως βουλευτές, διότι πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη το θέμα των θεμελιωνών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα από τα καθήκοντά μας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Ε, προκύπτει προφανώς από αυτή την ανταλλαγή απόψεων ότι το θέμα της ευρωπαϊκής ε, στρατηγικής ε, ασφάλειας ε, είναι ευρύτατο, αλλά ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλές διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Αυτό με οδηγεί πάρα πολύ ωραία στο να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Κάρμεν Ερμοσίν, η οποία θα μας δώσει, αν θέλετε, μια πρώτη εικόνα και θα εξαγάγει κάποια πρώτα συμπεράσματα. Κατόπιν τα τελικά συμπεράσματα θα τα δώσει η συνάδελφος, ε, η συμπρόεδρος, η κυρία Ίγκε Ντέιβιτσον. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο το καθήκον μου φυσικά. Ακούσαμε νομίζω περίπου 20 παρεμβάσεις, ε, οι οποίες θεωρώ ότι όλες ήταν επικοδομητικές, ενδιαφέρουσες και ουσιαστικά ανοίγουν νέες προτάσεις, νέες ιδέες και νέες μεθόδους. Όπως και να έχει, Θα κάνω μια πολύ γρήγορη αξιολόγηση και να πω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Θεωρώ ότι η πλειονότητα των παρεμβάσεων ε, ακολούθησαν αυτή την κατεύθυνση, τις δυνατότητες, τις προσδοκίες της νέας συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θα τεθεί σύντομα σε ισχύ και ε, η εξέλιξη των όσων θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Στοχόλμης ε, και με, με δύο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλουμε περισσότερα. Κάποιοι είπαν ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τις πολιτικές ασφαλείας, ε, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν τεθεί μέχρι τούδε, για να μπορέσουμε να τις δούμε και να τις συμπληρώσουμε να συμπληρώσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες οι οποίες είναι μεν εν εξελίξη αλλά όπως είπε και κάποιο, αν δεν είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι αν δεν δημιουργήσουμε νέες προδοκίε για αυτό το πρόγραμμα θα ε, καταλήξουμε σε λιγότερες απαιτήσει. Αυτή νομίζω λοιπόν είναι η άγουσα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό το οποίο ακούστηκε επανειλημμένος ε, νομίζω ότι ήταν το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και την προσαρμογή του στα νέα μέσα τα οποία ε, θα χρησιμοποιηθούν για να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης και η συνθήκη της Λισαβόνας και πιο συγκεκριμένα όλα όσα έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, τους παράνομους μετανάστες και το δικαίωμα του ασύλου. Στην ε, χώρα μου μόλις εγκρίναμε τις προηγούμενες ημέρες ε, μια νέα νομοθεσία για το άσυλο η οποία ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τις οδηγίες και ε, κάποιος είπε και λίγο πριν ε, αφορά και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι ερίζουν οι απόψεις στα θέματα του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι από τους προλαλήσαντες αναφέρθηκαν επίσης στην καταπολέμηση των ε, σοβαρών αδικημάτων, ε, την εμπορία ανθρώπων και επίσης θα πρέπει να υπάρχει πάντα ασφάλεια. Και υπάρχει και ένας κοινό παρονομαστής, ο οποίος νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη όταν μιλάμε για την ασφάλεια και είναι το θέμα της ισορροπίας και της συμβατότητας μεταξύ ασφάλειας και ελευθεριών την ασφάλεια των πολιτών και των ελευθεριών και τα μελωδών τους δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι όπως πολύ σωστά είπε ο κύριο Κοέλιο, δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια χωρίς ελευθερία, αλλά ούτε και ελευθερία χωρίς ασφάλεια ε, θα ήταν αντιπαραγωγικό να λείπουν και τα δύο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα όσα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, συστήματα πληροφόρησης, ποινικά συστήματα, δικαστικά συστήματα. Όλα αυτά είναι υπό τη σκέπη της διασφάλισης των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ε, ανθρώπων, τα οποία θα μας οδηγήσουν φυσικά ε, στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. Τίποτα άλλο, θα τα μελετήσω όλα, θα ε, λίγο αργότερα βέβαια σήμερα. Ευχαριστώ. Υπήρξε ένα πρόβλημα αρχικά με το μικρόφωνο. Νομίζω ότι η σύνοψη που μας έκανε η συγγήτρια η κυρία Ερμοσίν ήταν καταπληκτική δεδομένο το πόσο λίγο χρόνο είχε για να ανακεφαλαιώσει τις αδερές γραμμές της συζήτησης. Και εγώ παρόμοιες απόψεις έχω. Νομίζω ότι η τιμιγορία του, των ομιλητών για το πρόγραμμα της Στοχόλμης ήταν μάλλον θετική. Απλώς οι περισσότεροι ζήτησαν κάποιες πιο πρακτικές διατάξεις και μία πιο ενδελεχή αξιολόγηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα της Χάγης. Πολλές αποφάσεις ελήφθησαν και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρξε πάντα σωστή, αρκετή συμμόρφωση, σωστή εφαρμογή τους. Πολλοί τάσσονται υπέρ της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνδρομής, ακόμη και των κοινών ερευνών, αλλά και της ανάγκης ανταλλαγής ε, πληροφοριών ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική ασύλου, νομίζω ότι αναφέρθηκε και η ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών που φέρνουν την κύρια ευθύνη ε, για την πολιτική ασύλου, αλλά ταυτόχρονα και την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες που έχουν λόγους για τους οποίους αποφεύγουν τη χώρα τους. Φεύγουν μερικές φορές ακούσια για να γλιτώσουν από ανυπόφερες καταστάσεις. Η Σουηδία έχει δεχτεί πάρα πολλούς ετούντες άσυλο σε σχέση με τον πληθυσμό της και μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την φιλοξενία αυτή που δείξαμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης του εγκλήματος και της προάσπισης της ακαιρεότητας ή των ατομικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες είναι όλο και πιο δύσκολη και έθραυστη αυτή η ισορροπία. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο για μας, να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο ετοιμάτων. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά γιατί πιστεύω ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Και νομίζω ότι αύριο που θα γίνει νέα ανακεφαλαίωση της συζήτησης, ε, οι συγητές θα μπορέσουν με ακόμη καλύτερο και ευσύνοπτο τρόπο να, να, να αντικατοπτρίσουν αυτά που υπόθηκα. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.